Σταθεί μια ομάδα που λεγόταν MAG, δηλαδή βουλευτές κατά του καρκίνου. Νομίζω τώρα πως με τη νέα ομάδα θα δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην πρόληψη. Σας ευχαριστώ όλους και καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε κύριε Πέτερλε. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί. Περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η έκθεση της κυρίας Τόγια για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Η κυρία Τόγια έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Η έκθεση που συζητάμε σήμερα και θα ψηφιστεί αύριο αφορά την εφαρμογή του πακέτου 2020-2020 που είναι το πιο μακρόπνο σχέδιο της προηγούμενης θητείας. Αν μου πείτε τι πρέπει να περισσώσω από τα προηγούμενα πέντε χρόνια, θα ε, υπόψη αυτό το πακέτο 20-20-20. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ε, έγινε εντατική εργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε μία ανακοίνωση και μία σύσταση και την εργασία της Επιτροπής Ήτρε και άλλων με πολλές υποδείξεις, τροπολογίες και εμπλουτισμό της εργασίας μας. Νομίζω ότι υπάρχει διχογνωμία ως προς ένα σημείο και ελπίζω ότι με την αυριανή ψηφοφορία θα το ξεπεράσουμε. Πρόκειται για το δεσμευτικό χαρακτήρα που θέλουμε να αποδώσουμε σε αυτή την έκθεση ως προς το περιεχόμενο. Θα ήθελα όμως να πω ότι υπήρξε ομοφωνία γενικότερα. Οι τεχνολογίες ICT, οι τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας αποτελούν ένα πολύ σημαντικό τομέα που βαρύνει ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μιλάμε για 7% του εργατικού δυναμικού, του ευρωπαϊκού και 6% του ΑΕΠ. Άρα δεν είναι καθόλου αμεληταίο αν λάβουμε υπόψη την ε, παραγωγική οικονομία στα πλαίσια των ευρωπαϊκών συμφραζομένων. Αυτό που έχει σημασία είναι ο ουσιώδης ρόλος αυτής της ε, τεχνολογίας για να μεταβεί η οικονομία μας σε ένα ιδιαίτερα αναπτυξιακό πλαίσιο με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, άρα ε, λιγότερη μόλυνση για τις μελλοντικές γενναίες. Να περάσουμε σε πραγματικά γεγονότα, σε μια υλοποίηση ενός νέου τρόπου ζωής και κίνησης, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια βιομηχανική επανάσταση που θα χαρακτηρίζει την οικονομική και κοινωνική ζωή του μέλλοντος, όχι μόνο της δικής μας Υπήρου, αλλά και όλων των άλλων. Πώς μπορούν αυτές οι τεχνολογίες, το ITC, να μας βοηθήσει, αλλάζοντας τον ίδιο τομέα, το τομέα. Πιστεύω ότι έχει σημασία να εξεύρουμε μέσα επικοινωνίας και μικροηλεκτρονικής για να καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια και μπορούν να συνεισφέρουν και οι μεγάλοι τομεί των κτηρίων, των κατασκευών και των μεταφορών. Παίρνω τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου μία καλύτερη απόδοση των στόχων 20-20-20 θα μας οδηγούσαν σε μία μείωση γιατί οι μεταφορές αποτελούν το 27% της ενέργειας, το 40% αφορά τις κατασκευές, ε, σύστημα ψήξης θέρμανσης, άρα η μείωση αυτών των εκπομπών θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα υψηλή, με μεγάλη σημασία. Και τα πεδία εφαρμογής είναι πολύ μεγάλα και αφορούν πολλούς τομείς τραπεζικός τομέας, δημόσια διοίκηση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ούτω καθεξής, όπου μπορούμε να έχουμε εξοικονόμηση εκπομπών αλλά και χρόνου, να βελτιώσουμε δηλαδή την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την κοινωνική ζωή. Νομίζω όμως ότι ακόμα πιο σημαντικό θα ήταν αύριο να εγκρίνουμε το δεσμευτικό χαρακτήρα. Τα smart meters και τα, ε, οι ευφυείς πόλεις καθώς και τα ε, ευφυή ε, ηλεκτρικά δίκτυα μπορούν να διαδραματίσουν μεγάλο ρόλο. Ε, οι δήμαρχοι μίλησαν για μια συμφωνία μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων έτσι ώστε να υπάρχει ε, ουσιαστική ενεργειακή απόδοση και μεγαλύτερη και καλύτερη ε, ποιότητα ζωής. Τώρα περνάμε στο Catch the Eye. λόγο έχει η κυρία Μάκοβέη. Όχι. Ε, Είμαι σκιώδης εισηγήτρια στην έκθεση Κοτσολίνο εγώ στην ε, επόμενη, μεθεπόμενη. Ωραία, η κυρία Πασέσκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι τα ευρωπαϊκά ταμεία θα πρέπει να φτάσουν στον Ευρωπαίο πολίτη. Αν θέλουμε να μειώσουμε την ε, διαφθορά στα συστήματα δημόσιων προμηθειών, θα πρέπει να έχουμε ένα διαφανές σύστημα διαγωνισμών. Πιστεύω ότι η εφαρμογή νομοθετικών και θεσμικών μέτρων από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποθαρρύνουν την απάτη και στέφθηκαν από επιτυχία. Χρειαζόμαστε ε, χρηματοοικονομικό έλεγχο και μία αποτελεσματική καταπολέμηση των απατών στον τομέα του ΦΠΑ. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα για τη ρουμανική κυβέρνηση που έχει ένα ειδικό τμήμα για την καταπολέμηση διαφθοράς και απάτης και είμαστε σε άμεση επαφή με την όλα. Κύριε Μπασέσκου, αναφερθήκατε στο επόμενο σημείο, σε μια άλλη έκθεση. Εντάξει, εντάξει, τα είπατε, τα είπατε. Εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Προτρέξατε, αλλά δεν πειράσει. Το λόγο έχει η κυρία Τσικάου, η ακάματη θα ήθελα να χαιρετήσω τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου του 2010 που αναφέρεται στην ανάγκη αύξησης κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης. Και αυτό σχετίζεται με την χρήση των ε, τεχνολογιών επικοινωνίας, ε, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιήσουμε τα ευφύ δίκτυα. Όλα τα συστήματα που βασίζονται στις ε, τεχνολογίες πληροφορίας, και επικοινωνίας μπορούν να μειώσουν τις ενεργειακές ανάγκες κτηρίων μέχρι 60% και μπορούμε να φτάσουμε στο τομέα των μεταφορών στο 27%. Τα ηλεκτρικά δίκτυα επίσης θα πρέπει να μετατραπούν σε ευφύ δίκτυα και η ηλεκτρική ροή θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη εξαιτίας των ITC. Επίσης θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο μέσα στα πλαίσια του ευρυζωνικού. κυρία Μπασέσκου. Συγγνώμη, επειδή μας δώσατε σε μένα και την άλφο το λόγο ε, για να μιλήσουμε για την ε, καταπολέμηση της απάτης. Κάπου ακούστηκε η λέξη απάτη, εν πάση περιπτώσει. Και περάσαμε στο επόμενο θέμα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κανένα πρόβλημα, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει τη στήριξη και τις συστάσεις σας για την κινητοποίηση των τεχνολογικών πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και διαβάσαν προσεκτικά την έκθεση ΤΟΙΑ. Είναι σημαντικό να γνωρίσουμε τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο τομέας της πληροφορική στη μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου και να διασφαλίσουμε πώς θα γίνει πραγματικότητα αυτή η δυνατότητα. Εμείς σκοπεύουμε να δώσουμε προτεραιότητα στο θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα που θα υιοθετηθεί προσεχώς. Όπως αναφέρεται, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών μπορούν να βελτιώσουν την ενεργειακή αποτελεσματικότητα σε άλλους τομείς, όπως τα κτίρια, τις μεταφορές ιδιαίτερα. Επίσης, συμφωνούμε πως τα έξυπνα δίκτυα και οι έξυπνοι μετρητές είναι σημεία κλειδιά Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε εμπερός εμείς και τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές την ε, ανανεώσιμη δημιουργία ενέργειας και την αποτελεσματική χρήση αυτής. Ε, μέτρα λοιπόν τα οποία θα συμφωνήσει και η βιομηχανία είναι σημαντικά για να δούμε πώς θα βοηθήσουν οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Από την υιοθέτηση της, ε, ίσταση, της σχετικής τον Οκτώβριο του 2009, η Κομισιόν έχει αναλάβει μια σειρά δράσεων με ενδιαφερομένους για να την προωθήσει. Να αναφέρω κάποια πράγματα που αφορούν αυτά τα οποία είπατε στην εκθεσή σας το Φεβρουάριο του 2010. Το σχετικό φόρουμ ξεκίνησε. Το φόρουμ φέρνει σε επαφή ενώσεις βιομηχανίας πληροφορικής από τη ΣΥΠΑ, την Ιαπωνία και την Ένωση για να υπάρξει μια κοινή μέτρηση του αποτυπώματος του άνθρακα εντός του 2010. Επίσης το φόρουμ εξετάζει τη συνεισφορά που μπορεί να έχει ο κλάδος στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας άλλων κλάδων όπως τα κτίρια και οι μεταφορές. Μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν υπογράψει τον πράσινο ψηφιακό χάρτη με στόχο να μειώσουν κατά 30% έως το 2020 το ψηφιακό τους αποτύπωμα και να έχουν πέντε μεγάλης κλίμακας έργα μέχρι το 2015. Ο συνολικός αριθμός των πόλεων έχει αυξηθεί σε 21. Επίσης σημαντικά είναι τα ζητήματα της λιανικής αγοράς ενέργειας, καθώς η αγορά πηγαίνει πιο κοντά στους καταναλωτές με τους έξυπνους μετρητές και τα έξυπνα δίκτυα. Η συνεργασία με τη σχετική ομάδα της Κομισιόν επίσης προχωρά έτσι ώστε να συμβουλεύσει την Κομισιόν για το ρυθμιστικό πλαίσιο και να συντονιστούν τα πρώτα βήματα για τα έξυπνα δίκτυα σύμφωνα με το τρίτο ενεργειακό πακέτο. Αναμένουμε συστάσεις μέχρι το τέλος του 2011. Τελειώνω λέγοντας πως η Κομισιόν θα συνεισφέρει βεβαίως στην επίτευξη των στοχων 2020 2020-2020 όπως θα όρισε το Συμβούλιο και βεβαίως πληροφορική έχει σημαντικό ρόλο να παίξει. Σας ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας με την έκθεσή σας και αναμένουμε να συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε πώς θα έχουμε τις κατάλληλες πολιτικές. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η έκθεση αυτή θα ψηφιστεί αύριο. Τελευταίο σημείο για σήμερα είναι η έκθεση